πρακτικών. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσης διάταξης, προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020. Μία είναι η συντάκτηρα της προφορικής ερώτησης, η κυρία Ουσκοκ την οποία και δίνω το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη πλήττεται ε, από την ε, κρίση ε, και φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την αγορά εργασίας γίνονται πιο επικίνδυνες οι συνθήκες πλέον στην αγορά εργασίας. Ε, χρειαζόμαστε ε, νομοθεσία ισχυρή η οποία θα διέπει την εργασία και που θα αφορά όχι μόνο όσους ε, εργάζονται και που είναι στις εταιρείες αλλά και τις ίδιες τις εταιρείες. Σύμφωνα με μελέτες, εάν μία μία ε, εταιρεία επενδύσει 10 ευρώ στην προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων, τότε ε, θα τις επιστραφεί στο διπλάσιο ε, το ποσό αυτό. Θα πρέπει να δημιουργηθεί επίσης ένα ίσο επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στρέβλωση της αγοράς λόγω των πολλών και διαφορετικών κανόνων. Τα πρότυπα πρέπει να είναι υψηλά, αλλά και η απλούστευση ε, να είναι μεγάλη. Θα πρέπει να μειωθεί ε, η γραφειοκρατία ε, και θα πρέπει να λαμβάνονται, θα πρέπει η νομοθεσία να είναι πιο απλή έτσι ώστε αποτελεσματικά να προστατευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί έτσι όπως έχει η κατάσταση δημιουργούνται προβλήματα και για τους εργαζόμενους και για, τις, για τους εργοδότες. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίε βεβαίως μπορεί να μην καταλαβαίνουν τέτοιου είδους προβλήματα αλλά για μια μικρή επιχείρηση ε, πρέπει, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος να είναι στην θέση του δηλαδή ε, να μην αρρωσταίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα γιατί η κάθε θέση εργασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική όλοι θα πρέπει να έχουν ε, δικαίωμα σε καλό εργασιακό περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα ε, το οποίο μπορεί να εξαχθεί. Ναι, Βεβαίω, το Κοινοβούλιο έχει συζητήσει πολλές φορές τα θέματα αυτά. Περισσότερο από το 90% των ε, εργοδοτών ε, από της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά τον χώρο εργασίας. Γιατί αυτοί οι κανόνες αφορούν μονάχα τις πολύ μεγάλες επιχειρήσει είναι εξαιρετικά σημαντικό τώρα στην αρχή αυτής της ε, κοινοβουλευτικής ε, θυσίας θητείας ε, να ε, μπορέσουμε να πάρουμε τα σωστά μέτρα έτσι ώστε ε, οι κανόνες να είναι σωστοί και να εφαρμοστούν κυρίως σωστά. Ακούμε για νέα προγράμματα, ακούμε για νέες πολιτικές διαχείρισης, για βοήθεια σε μικρές επιχειρήσεις, κατάρτιση ε, ε, κατάρτιση ακόμα και των ε, συνδικάτων έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα εργασιακά περιβάλλοντα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η επιδίνωση του εργασιακού περιβάλλοντος που διαπιστώνεται στις περισσότερες θέσεις εργασίας. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων ε, σε ε, ατυχήματα αλλά κυρίως ε, και σε καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες καθώς επίσης οτιδήποτε σχετίζεται με μειοσκελετικά αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού θα λειτουργούν σωστά και ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε να έχουμε μια κοινωνία ισχυρή που θα εργάζεται εργάζεται με σωστές συνθήκες. Ευχαριστώ. Η κυρία Επίτροπος, παρακαλώ. Ε, ναι, Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Απασχόλησης, μέλη του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στεναρά προσιλωμένη στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και υγείας και υγιεινής στην εργασία. Η νέα στρατηγική και το πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εγκρίθηκε τον Ιούνιο αντανακλά ακριβώ αυτές τις δεσμεύσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ μεγάλο σώμα νομοθεσίας ήδη ε, περί αυτών. Το νέο στρατηγικό μας πλαίσιο έρχεται να συμπληρώσει το ε, κεκτημένο ε, δίνοντας μια ε, συνολική κουλτούρα πρόληψης και δίνει και ένα πλαίσιο για να συντονίζονται οι εθνικές πολιτικές και να βελτιώνεται η υλοποίησή τους. Το πλαίσιο εντοπίζει τρεις βασικές προκλήσεις. Πρώτο, βελτίωση της εφαρμογής της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και της αντίστοιχης νομοθεσίας ιδιαίτερα με ενίσχυση της δυνατότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων να ε, υιοθετούν ε, μέτρα πρόληψης αποτελεσματικά. Το δεύτερο είναι να ε, βελτιωθεί η πρόληψη των επαγγελματικών νόσων με αντιμετώπιση των νέων αναδυόμενων κινδύνων και το τρίτο είναι αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής και της γύρασης του εργαζομένου πληθυσμού. Ε, και δυναμικού. Για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται ενεργή συμμετοχή όλων των ενεχομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με τα κράτη-μέλη, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγιεινής Συνεργασία, ε, με την Τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγιεινή Συνεργασία, καθώς επίσης ε, και την Επιτροπή Επιθεωρητών εργασία, υψηλού επίπεδου για να είναι σωστή η υλοποίηση των υφισταμένων κανόνων. Και οι δύο επιτροπές και ο οργανισμός αναθεωρούν τα προγράμματα εργασίας ε, υπό το φως του νέου στρατηγικού πλαισίου. Θα συνεχίσω εγώ να ενέχω και τους κοινωνικούς εταίρους αυτή την προσπάθεια μέσω του κλαδικού διαλόγου που έχουμε όταν αυτό χρειάζεται. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμερής για την Ασφάλεια και την Υγεία Συνεργασία βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βελτιωθεί καλύτερα η παρακολούθηση της υλοποίησης. Ε, σημείωσα στην προφορική σας ερώτηση το αίτημα να εισαχθούν ειδικοί δείκτες ε, σε σχέση με όλα αυτά. Ε, διάφορα μέτρα ήδη εφαρμόζονται, όπως είναι η online εκτίμηση κινδυνού διαδραστική που έχει εκπονήσει ο οργανισμός και ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης επιθεωρητών εργασίας μια μελέτη για τη βελτίωση των επιθερήσεων εργασία σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα πάντα της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία ε, είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή και στο στάδιο της εκπόνησης. Ε, υπάρχουν ε, ήδη κανόνες και οδηγεί βέλτιση πρακτική, φιλικές προς το χρήστη πάντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει και τι πάρα πολύ μικρέ. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα το νέο στρατηγικό πλαίσιο έχει ένα νέο στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας στην εργασία. Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αρχίσει μια ε, εκ των υστέρων αναθεώρηση και έλεγχο 24 οδηγιών ε, με το αποτέλεσμα να αναμένεται στα τέλη του 2015. Επιπλέον το στρατηγικό πλαίσιο τονίζει την ανάγκη ε, να δούμε τον αντίκτυπο στην σωματική και ψυχική υγεία ε, στον χώρο εργασίας και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό. Το πλαίσιο επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι στατιστικές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγιεινή εργασία και να δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων. Οι στατιστικές είναι χρήσιμες και κρίσιμες για να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην εργασία και οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Συνεχίζεται η αξιολόγηση ε, των αντιστοίχων οδηγιών και τα αποτελέσματα θα είναι αποφασιστικά για να δούμε αν χρειάζεται νέα νομοθεσία, ενδεχομένω νέε νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Η ασφάλεια και η υγιεινή συνεργασία και η αντίστοιχη νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται πάντα σε στοιχεία και όποια νέα πρόταση θα ε, βασιστεί σε μια βαθιά μελέτη αντικτύπου. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Ο κύριο Μπέκερ έχει το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κατά πλειοψηφία 46 υπέρ 1 κατά και μία αποχή στην Επιτροπή Απασχόλησης αποφασίσαμε την ε, προφορική ερώτηση αυτή και ομόφωνα έχουμε ε, διατρανώσει ότι δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι με την κατάσταση των πραγμάτων ως προς τις προτεραιότητες για τα επόμενα έτη. Πάρα πολύ συχνά έχουμε πολύ βαριές ασθένειες που συνδέονται με εργατικά ατυχήματα και με προβλήματα επαγγελματική ιατρικής που έχει και υψηλό κόστος αυτό για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ε, απουσία από την εργασία και χάνουν χρήματα και εισόδημα και εργαζόμενοι και εργοδότες. Από τα λεγόμενα σας κυρία Επίτροπε, ε, κατανοώ ότι τα έχετε καταλάβει κι εσείς όλα αυτά, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αλλιώς δεν θα είχατε προχωρήσει σε αυτή την προσπάθεια. Και με ικανοποίηση διαπιστώνω ε, ότι επιλέγετε μια σφαιρική αντιμετώπιση και την προτιμάτε. Ωραία. Αλλά χρειαζόμαστε στόχους πιο συγκεκριμένους και προθεσμίες πιο δεσμευτικές. Ωραίο το στρατηγικό πλαίσιο, αλλά λείπουν όλα αυτά και θα πρέπει να δούμε και την παρακολούθηση των κινδύνων ε, για την υγεία και να δούμε και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος και των επαγγελματικών ασθενειών. Αυτά ε, δεν έχουν λυθεί ακόμα. Γενικά πιστεύω ότι δεν είμαστε ακόμα στο τέλος του δρόμου και θα χαιρόμουν εάν σε μελλοντική μας ε, συνεργασία μας σας σε ένα απότερο στάδιο είχαμε την ευκαιρία πολύ συγκεκριμένα να μιλήσουμε για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Στάινρουκ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε αρκετά αργά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2011 είχε ζητήσει μια στρατηγική που θα συνεχίζει την προηγούμενη. Και ομολογώ ότι αυτό που μας έχετε φέρει δεν είναι πραγματική στρατηγική, το είπε και ο συνάδελφος. Λείπουν συγκεκριμένες προτάσεις, βελτίωση, χρονικό περιθώριο, πλαίσιο, στόχοι και πάντα έχουμε νέες ε, προκλήσεις, αλλάζει η τεχνολογία, έχουμε και νέους τύπους εργασίας, νέες ασθένειες. Ένα παράδειγμα μόνο να σας δώσω. Πάνω από 80% των ε, καταθλίψεων είναι κατά τη διάρκεια του εργατικού βίου και ένας στου δέκα εργαζομένους ε, λείπει από την εργασία του για λόγου κατάθλιψης. Χρειάζονται προγράμματα πρόληψη, ασφάλεια και προστασία τη υγιεινής στην εργασία. Πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά. Εμεί είμαστε νομοθέτε και είμαστε υποχρεωμένοι ε, να εξασφαλίζουμε ένα υγιή εργασιακό βίο. Και ανησυχώ για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για λόγους ε, μη γραφειοκρατία εξαιρούνται ενδεχομένω από ορισμένε ρυθμίσει. Υποτίθεται ότι αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα. Αλλά αυτό που αποσιωπάτε είναι ότι ε, το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Δεν το πληρώνει η εταιρεία, αλλά το πληρώνει το γενικό σύνολο ε, και με τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα ε, συστήματα τα ασφαλιστικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόληψη και η εφαρμογή να γίνεται καλύτερα και καλύτερα από το να αναφέρουμε γενικά κάποιους κινδύνους. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μακιντάιρ. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την αναθεώρηση, γιατί χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ασφάλειας και υγείας στην εργασία, γιατί αλλάζουν ε, οι μορφές εργασίας και έχουμε νέους ή αναδυόμενους κινδύνους. Κάθε αναθεώρηση όμως ε, θα πρέπει να αναγκαλίζεται τις αρχές του εφνομοθετήν. Χρειαζόμαστε λοιπόν νομοθετικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία. Δεν θέλω μέτρα που θα μειώνουν την, ε, ή θα υποβαθμίζουν την υγεία. Θέλουμε να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε την ασφάλεια και την υγεία, κάτι που δεν ισχύει με τι τελευταίε προτάσει. Θα πρέπει να μειώσουμε την περιπλοκότητα τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία γιατί μόνο έτσι θα αυξήσουμε τη συμμόρφωση, θα υλοποιήσουμε τους στόχους για ενισχυμένη ασφάλεια και υγεία στην εργασία και θα μειώσουμε και το γραφειοκρατικό φόρτο για τις ε, επιχειρήσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι επιθεωρήσεις ασφάλειας και υγείας θα πρέπει να επικεντρώνονται στο τι συμβαίνει πραγματικά στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο αντί να επικεντρώνονται στην ε, σχολαστική ε, έρευνα των εγγράφων. Θα ήθελα να ε, μειώσουμε την γραφειοκρατία και να ε, απλουστεύσουμε την νομοθεσία. Επίσης, ε, η τεκμηρίωση για την αξιολόγηση κινδύνου στις μικρές επιχειρήσεις σε τομείς χαμηλού κινδύνου θα πρέπει και αυτή να απλουστευτεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την απάντηση και την απόκριση της. Ας μην ξεχνούμε ότι κάθε χρόνο πάνω από 4.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι εργαζόμενοι είναι θύματα εργατικών ατυχημάτων και πρέπει να απουσιάσουν τουλάχιστον τρει μέρε από την εργασία του. Μιλάμε για εντυπωσιακά ποσά. Μιλάτε για 11 ανθρώπου τη μέρα που χάνουν τη ζωή του καθημερινά και πάνω από 800 που τραυματίζονται. Γι' αυτό λοιπόν θέσαμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα που δεν περιμένουν να απαντηθούν όλα φυσικά, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε ορισμένα τουλάχιστον. Όταν μιλούμε για μετρήσιμους στόχους που θα διορθώσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις περιοδικές ε, αξιολογήσεις, θα ήθελα να ρωτήσω αν όντως σημειώθηκε πρόοδος στη βελτίωση της κάλυψης των στατιστικών πληροφοριών, την ε, αξιοπιστία τους, τη συγκρισιμότητά τους, την ε, επίκαιρη και έγκαιρη υποβολή τους. Υπάρχει πρόοδος στα σημεία αυτά. Επίσης, τι δράσεις υιοθετήθηκαν για να προαχθεί η ανταλλαγή των πρακτικών. Για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίσως θα μπορούσαν να στηριχτούν, να βοηθηθούν ή να λάβουν συμβουλές από μεγαλύτερε εταιρείε στην αλυσίδα αγοραστή πολιτή. Επίσης υπάρχουν κάποιε της πρωτοβουλίες και μιλήσατε για τη χρήση και έκδοση εγχειριδίων φιλικών προ το χρήστη. Μπορείτε να μα αναπτύξετε κάπω πιο διεξοδικά αυτό το σημείο. Επίσης, ε, αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες με βάση το φύλλο και την ηλικία. Πολύ σημαντικά αυτά τα αναλυτικά στοιχεία για το φύλλο και την ε, ηλικία. Θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε μια καλύτερη ιδέα για το τι συμβαίνει. Τέλος, ε, σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου μάθαμε ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι το άγχος είναι ο μείζον κίνδυνος επαγγελματικός. 53% των εργαζομένων θεωρούν το άγχος ως κύριο υπέτειο. Και μάλιστα το Ίδρυμα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία έχει ξεκινήσει εκστρατεία ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά. Αλλά μια και είναι τόσο υψηλό ο κίνδυνο ε, του άγχου στον εργασιακό χώρο, δεν πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε πιο άμεση δράση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ποιες είναι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν προτάσεις για να προωθηθεί η ενεργέ περιβάλλον και μία ψυχική ε, ε, ευεξία στον εργασιακό χώρο. Επίσης, ε, σε ό,τι φορά την οδηγία για τις μειοσκελετικέ ασθένειες, δυστυχώς κατέπεσε στο Συμβούλιο η οδηγία αυτή, εκεί να βάγισε. Και πάλι σα παραπέμπω στη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου που λέει ότι ένα στου τέσσερι εργαζόμενους θεωρεί ότι η εργονομική κίνδυνη είναι πολύ σημαντική. Και ίσω δεν χρειάζεται εδώ οδηγία, αλλά κάποια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπόιλαν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε το θέμα τη ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο και χαίρομαι για την δεδηλωμένη πρόθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων. Δεν μπορούμε από τη μια όμω να έχουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, όταν από την άλλη υιοθετούμε πολιτικέ που οδηγούν σε επισφαλεί και ανασφαλεί εργασιακού όρου. Δυστυχώ αυτή είναι η κανόνα, ο κανόνα και στην Ιρλανδία 46% αύξηση των συνθηκών αυτών είχαμε και υποαπασχολούμενος εργαζόμενος Και μάλιστα ε, για τους ε, κοινωνικο-οικονομικούς κινδύνους δεν θα πρέπει να υποτιμούνται και η πίεση και το άγχος από τις ε, υπερβολικές υπερορίες οδηγούν στις απουσίες και επίσης οι χαμηλοί μισθοί έχουν, αρνητικό αποτέλεσμα, έχουν αρνητική επιρροή στην πρόσβαση σε θρεπτικές τροφές και σε σωστή υγειονομική περίθαλψη για τους εργαζόμενους. Αν λοιπόν κοπτόμαστε για την ασφάλεια και την υγεία, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τους επισφαλείς όρους απασχόλησης και τους χαμηλούς μισθούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλαμε να βελτιώσουμε την υγεία των ε, Ευρωπαίων και είχαμε φιλοδοξου στόχου. Ε, το 2011 αυτό πριν τρία χρόνια και σήμερα για το 2014-2020 το πλαίσιο δηλαδή τη Κομισιόν ε, είμαστε τέτοιοι φωτός. Ε, Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που υφίστανται ατυχήματα και νόσους που σχετίζονται με, τις, ε, με την εργασία. Είναι ηθικό σφάλμα να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στους ανθρώπους που υποφέρουν στην εργασία και όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά στις επιχειρήσεις μας και στο σύστημα υγείου μας. Ποιους δείκτες σκοπεύετε να θέσετε σε ό,τι αφορά ε, το θέμα της ανισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία και πότε θα εμπλέξετε τους κοινωνικούς ιδιωτικού εταίρου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε το 2006. Πότε θα δώσετε ορισμό ε, για τα επαγγελματικά ατυχήματα και τι νόσου, ε, το πλαίσιο που έχετε δεν ανταποκρίνεται και ο κύριος Γιούνκερ λέει συχνά ότι η Κομισιόν ε, έχει, τις, τελευταία τη δυνατότητα, εγώ θα λέγω την τελευταία ευκαιρία της Κομισιόν να ανταποκριθεί γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν πλέον να χάνουν τη ζωή τους. Ευχαριστώ κύριο Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Οι τελευταίε εκτίμησει τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την έρευνα για τον καρκίνο δείχνει ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε κάθε χρόνο αρρωσταίνουν με καρκίνο. Το 8% αυτών των πολιτών αρρωσταίνει λόγω εκθέσεω επαγγελματική εκθέσεω. Αν στι επαγγελματικέ εκθέσει έχουμε την έκθεση στον αμίαντο και στι ίνε. Το 56% των περιπτώσεων του, μεσοθυ... του πλευρικού μεσοθυλιώματο, 43% τη αμοιαντιώσει προέρχονται στην Ευρώπη, όπου έχουμε μόνο το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και αν πηγαίνουν άσχημα τα πράγματα για την έκθεση στι ίνε του αμοιάντου, σίγουρα πάει χειρότερα όσον αφορά τον πετρελοχημικό τομέα όσον αφορά τη χαλιβουργία, ε, τα τσιμεντουργία. Θα, εγκαταλ... θα, θα τα εξαλείψουμε αυτό, αυτή την ασχήμια. Ε, αυτά είναι θέματα που περιμένουν τα κράτη-μέλη τα λύσουν, μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα κράτη-μέλη, όπω και η Ιταλία, έχουμε και το σκάδιο έτερνη για να σωθεί μόνο ένας πολιτικός. Χιλιάδες ε, πολίτες δεν ε, διέχτηκαν δικαιοσύνη. Να θέσουμε τέρμα σε αυτή την ασχήμια. Señor Mann. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σημαντικό όσον αφορά το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε πως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι απλά κάτι που θα πρέπει να επιβάλλεται. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν πως η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα και την απόδοσή τους, άρα και την ανάπτυξη των εταιριών τους. Ένας παράγοντας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το θέμα που συζητάμε είναι η πρόληψη εκτός από τα επαγγελματικά ατυχήματα που προκαλούνται συχνά από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια των μέτρων προστασίας αναφέρομαι και στις επαγγελματικές ασθένειες ένα πεδίο σχετικά παραμελημένο. πολλοί εργαζόμενοι προσβάλλονται από διάφορες μορφές καρκίνου δερματικές παθήσεις μυοσκελετικά προβλήματα και άλλες ασθένειες εξαιτίας των συνθηκών εργασίας και των υλικών με τα οποία έρχονται σε επαφή. όμως πώς μπορεί να υπάρξει πρόληψη όταν λόγω της κρίσης και της πολιτικής τη λιτότητα, χώρες όπως η ελλάδα βιώνουν μια πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας θα αναφέρω μόνο πως για μια απλή εξέταση ένας ασθενής στην ελλάδα έχει μέσο χρόνο αναμονής έξι μηνών. καταλαβαίνετε λοιπόν πως κάτω από αυτές τις συνθήκες το να μιλάμε για πρόληψη είναι εκτός πραγματικότητας. η πρόληψη σώζει ζωές αλλά μερικούς ενδιαφέρει στην πραγματικότητα μόνο η ευημερία των αριθμών και όχι των λαών. με την επαγγελματική της λιτότητα των μνημονίων και τις επιταγές της τρόικα οι εργαζόμενοι απλά αφήνονται στην τύχη τους. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαν έχει το λόγο. Οι συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε ότι θέλουν να βελτιωθούν. Ε, θέλουμε να έχουμε και την ηγετική θέση στο θέμα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Ε, πράγματι, στην περίπτωση αυτή χρειαζόμαστε ε, περισσότερη Ευρώπη. Τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν σιω ε, ατυχήματα στην Ευρώπη. Για την εξομοίωση των συνθηκών εργασίας στις διάφορες χώρες, η οδηγία πλαίσιο ήταν ε, σημαντικότητα σε μια επανάσταση. Τώρα χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο και εμεί στην Επιτροπή απασχόληση είπαμε ότι χρειαζόμαστε, θα πρέπει να διατυπώσουμε νέους στόχους και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους στις ε, μικρές επιχειρήσεις εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη επέμβασης γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου οι διατάξεις ασφαλείας δεν ε, τηρούνται κυρίως λόγω του υψηλού κόστους. Εγώ δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας ε, περισσότερης γραφειοκρατίας αλλά θα πρέπει να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας ούτως ώστε να προσαρμοστούν και οι νομικές διατάξεις και οι μικρές τις επιχειρήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της ε, αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας, ούτως ώστε να μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σάιμον. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν θέλω να το πω, αλλά κανά έκανε αυτό που έκανε το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή είπε καλά λόγια, έκανε τους σωστούς ήχους, αλλά παρουσίασε ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι στρατηγικό και δεν είναι καν πλαίσιο. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Πρόεδρε, ε, δεν περιέχει τίποτα, είναι κενό περιεχομένου. Πού είναι τα καρκινογόνα και σχετική διάταξη. Ο καρκίνος ξέρουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος των ανθρώπων στον χώρο εργασία και δεν βρίσκεται σε αυτό το υποτιθέμενο στατικικό πλαίσιο. Πού είναι ο αμίαντος που σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ε, το χρόνο. Πού είναι σε αυτό το υποτιθέμενο στρατηγικό ούτω αποκαλούμενο πλαίσιο. Τι γίνεται με το να έχουμε μαύρη λίστα. Ε, μπαίνουν σε μαύρη λίστα, 5.000 μπήκαν κάποιοι σε μαύρο κατάλογο, κάποιοι άνθρωποι σε εργοτάξια γιατί μίλησαν για την υγεία και την ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πού είναι η πρόβλεψη σε αυτό το στατικικό μη πλαίσιο. Τι γίνεται με την σωμάτωση ε, του καταλόγου με τις ε, ασθένειες ε, στον τόπο εργασίας που μπορεί να χρησιμοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Επίτροπος ε, είναι ειλικρινής στα θερμά της λόγια, το πιστεύω αυτό και στους ήχους τους ευ, ευμενείς που λέει, αλλά θέλουμε δράση για να κάνουμε τη διαφορά. Διαφορετικά ουσιαστικά είναι ένα παραπέτασμα καπνού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκυρίκια δεν είναι εδώ, δεν φαίνεται να είναι στην έδρα του. Από φαίνεται λείπει. Επομένως, να περάσουμε στην κυρία Ντορνάνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελούν το πυλώνα των επιχειρήσεων και τη ευημερία των μισθωτών. Καθώς πολλαπλασιάζονται οι τεχνικέ και έχουμε εμφάνιση νέων επαγγελματικών κινδύνων, τώρα οι ρυθμιστικές απαιτήσει θα πρέπει να διατηρηθούν. Η κρίση που περνάμε και που θα υποστούμε λόγω ενός οικονομικού έφερας του περιβάλλοντος είναι η βάρος της πρόληψης και στην επαγγελματική ασφάλεια εντός των επιχειρήσεων. Βέβαια είναι κάτι πανηρό, αλλά είναι απαραίτητο. Ας μην, κάνουμε, ας μην απατώμαστε. Η Ευρωπαϊκή, λύση δεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η λύση. Η Κομισιόν είναι υπερφιλελεύθερη και δεν μπορεί να υπερασπίσει την επαγγελματική ασφαλή και υγεία και ε, οι τεχνοκράτες ε, στις πολυεθνικές ονειφέρονται μια μεγάλη ελευθερία αγορά εργασίας στην Ευρώπη εις βάρος των κανόνων που θα υπερασπίζουν τους εργαζομένους. Είμαστε σε επιφυλακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι η γιατριά, δεν είναι η ίαση, αλλά η νόσος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ρολάν, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ναι. Ε, θα πρέπει να, να αναγνωρίσουμε τις ε, ε, τα προβλήματα. Ε, έγινε αναφορά στους αριθμούς. Πράγματι, κάθε μέρα έχουμε 11 νεκρούς στην εργασία. Κάθε μέρα είναι πάνω από 8.000 άτομα πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που μιλώ, 8 εργαζόμενοι θα πάθουν ε, ε, βαριά ατυχήματα στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι ανθρώπινο δράμα, αλλά έχει και έναν οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, έναν αντίκτυπο στην, στην ασφάλεια. Ε, πράγματι το πρόγραμμα αυτό διέπεται από πολιτική βούληση, αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε στις προθέσεις. Χρειάζεται να έχουμε στόχους ε, μετρήσιμους και κυρίως θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη, σε συνεχή δράση, η οποία να, να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε τα μέσα στα, για την ε, διενέργεια των ελέγχων και των επιθερήσεων. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία της κατάρτισης ούτως ώστε να υπάρχουν ε, νέα προϊόντα και νέες δεξιότητες. Κομισιόν ε, θα πρέπει να συνδράμει τους εργαζόμενους. Και τέλος, ε, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι αναγκαίο να απλουστευτούν επίσης οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει θέτοντα σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των μισθωτών εργαζομένων. Η υγεία και η ζωή τους δεν είναι δυνατόν να έχει ένα τίμημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιονγκέριος, παρακαλώ. Κυρία Επίτροπε, είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχουν λιγότεροι κανόνες για τις επιχειρήσεις, αλλά οι σωστές συνθήκες εργασίας υπερέχουν όλων των άλλων συμφερόντων. Ελπίζω ότι στην εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου θα κατορθώσετε να κάνετε την Ευρώπη τόπο όπου οι εργαζόμενοι ε, έχουν ένα καλό περιβάλλον. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι είχαμε αύξηση σειράς νέων μορφών εργασίας, ευέλικτη εργασία, ε, άνθρωποι που εργάζονται υπό συνθήκες εντελώς αβέβαιες και πρόσκαιρες, χωρίς καμία βεβαιότητα και χωρίς να διαθέτουν την ίδια προστασία όπως οι άλλοι εργαζόμενοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στοχευμένη προσέγγιση για αυτά τα άτομα, θα προβλέψει τα αναγκαία χέγγια για την ασφάλειά τους και για την υγεία τους στον τόπο εργασίας. Επίσης, υπάρχουν επιχειρηματίες που είναι εκτός του πλαισίου αυτού, όπως είναι στετιωτικοί ή αστυνομικοί, δεν έχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας. Εξού και ερώτησή μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για αυτά τα άτομα που ασχολούνται με τη δική μας ασφάλεια. Θα μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια εχέγγυα προστασία στον τόπο εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, για ένα λεπτό επόμενος ο και ο ευρωπαϊκή ένωση στον καπιταλισμό υγεία ασφάλεια ζωή των εργαζόμενων θεωρούνται κόστος και θυσιάζονται στα κέρδη για τα κέρδη. η νομοθεσία χαλαρώνει ελεγκτικές υπηρεσίες καταργούνται εργοδότες αθωώνονται για εργατικά ατυχήματα δολοφονίες εργατών που εκβιάζονται να σιωπούν για συνθήκες εργασία και ατυχήματα επιβαρύνονται για νοσηλεία και αποκατάσταση οι ίδιοι ζουν με αναπηρικά επιδόματα κοροϊδία εκατοντάδες δολοφονημένοι ανάπηροι εργάτες σε ναυπηγεία εργοστάσια μεταφορές στην ελλάδα έγκυες απειλούνται με απόλυση για να διακόψουν την κοίηση χιλιάδες πάσχουν από επαγγελματικές ασθένειες μετανάστες ζουν και εργάζονται σε άθλιες συνθήκες εκατοντάδες χιλιάδες πεθαίνουν στην ένωση από επαγγελματικές ασθένειες και είναι χιλιάδες τα θανατηφόρα ατυχήματα κάθε χρόνο. ασφάλεια ζωή υγεία των εργαζόμενων είναι πρώτη προτεραιότητα για το εργατικό κίνημα και τους κομμουνιστές που απαιτούν αυστηρή νομοθεσία προληπτικών μέτρων αποκατάσταση αναπήρων και ασθενών από επαγγελματικές ασθένειες και αποκλειστική επιβάρυνση κράτους και αποδοσία, ποινές στους υπεύθυνους και ικανοποιητικές συντάξεις στις οικογένειες των θυμάτων. Το θέμα που συζητούμε έχει ε, συζητηθεί πάρα πολύ και στη δική μου χώρα, σε διάφορους ε, τομείς, στην οικονομία, στον πολιτισμό. Είχαμε διάφορες ε, περίεργες υποθέσεις και είχαμε και το θέμα του αμίαντου. Είναι πραγματική μάστιγα και πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη στη χώρα μου. Η Ευρώπη είναι μια κοινότητα με μια πολύ προηγμένη νομοθεσία στο θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας, όμως δυστυχώς ε, αυτή η καλή νομοθεσία ε, στις χώρες γίνεται κάτι τυπικό και τεχνοκρατικό. Πώς ε, λοιπόν θα το αλλάξουμε αυτό. Ένας ε, νομικός στην Ιταλία, ο Μαρκο έχασε τη ζωή του για αυτά τα θέματα και έλεγε ότι πρώτα πρέπει να θέτουμε τους στόχους ε, και όχι τους κανόνες, τους σκοπούς. Ποιος είναι, ο σκοπός μας, κατάρτιση και ενημέρωση, αλλά όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των νέων οι οποίοι πρόκειται να μπουν στην αγορά εργασίας πρέπει να συνειδητοποιούν τι σημαίνει μια καλή δουλειά, πώς επιλέγεται κάτι τέτοιο και αν δεν μπορούν να την επιλέξουν, πώς την υπερασπίζουν και ε, με ποια αξιοπρέπεια. Αλλά θέλουμε και μια προσέγγιση να μην θεωρείται επικίνδυνος ο εργοδότης. Ε, εμείς ε, πιστεύουμε ότι μια όριμη οικονομία και τεχνολογικά προηγμένη θα ευνοήσει την ασφάλεια στην εργασία. Ευχαριστώ. Μπλινκεβίτσιτε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ ότι η πρόληψη του κινδύνου και η εφαρμογή των πολιτικών επαγγελματική υγείας και ασφάλεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Όμως ε, δεν μιλάμε εδώ για μία αυτόματη συσκευή, για μία μηχανή. Αυτό το νέο στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να στοχεύει στους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά και όλο ένα και περισσότερο καθώς ε, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Επομένως, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Οι εργοδότες θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις αλλαγές και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ε, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων. μην ξεχνούμε ότι ο επαγγελματικό κίνδυνος που προβλέπεται για τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους διαφέρει από αυτό για τους νέους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ε, ότι θα έχουμε τα κατάλληλα μέτρα στον επαγγελματικό τομέα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Παραδείγματος ε, χάρη αναφέρομαι στην ε, παρενόχληση των εργαζομένων ε, αν πρόκειται να τους απολύσουν, δηλαδή σε περίοδους κρίσης υπονοώντας ότι υπάρχουν άλλοι έτοιμοι να πάρουν τη θέση τους. Και πολύ λίγη σημασία δίνουμε στο άγχος που σχετίζεται με τη δουλειά. Όλα αυτά τα θέματα θα γίνουν ακόμη και πιο σημαντικά. Δεν μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι με τον ίδιο ρυθμό να προσαρμοστούν στις αλλαγές και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο στην ε, ψυχική και σωματική τους υγεία. Ευχαριστώ και θα ήθελα να παρατρύνω την Κομισιόν και διακόπτετε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο ο Πάπας έκανε έναν εμπνευσμένο λόγο και στο λόγο αυτό αναφέρθηκε κυρίως στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και ο καλύτερος τρόπος να δώσει κάποιον την αξιοπρέπεια είναι να του δώσει απασχόληση. Βελτιώνει την αυτοπεποίθησή τους και τους δίνει και ένα σκοπό. Δεν έχει νόημα όμως να δίνει κανείς σε κάποιον απασχόληση αν δεν είναι ασφαλής κανείς σε αυτή τη δουλειά. Και είναι σαφές ότι αυτό δεν συμβαίνει σε πολλά μέρη της ε, Ευρώπης και εδώ και λίγο καιρό ο Πρωθυπουργό της Λετωνίας είχε προβλήματα λόγω μιας καταστροφής που συνέβη στη χώρα. Και αυτό δείχνει ότι πάντα ελοχεύουν κίνδυνοι. Η Μαρία Χάρκεν το υποστήριξε το θέμα αυτό, τη θέση αυτή με στατιστικά στοιχεία. Πόσοι τραυματίζονται στον τόπο εργασία και είναι φρικτά, είναι τρομακτικά τα στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επεξεργαστούμε σωστά αυτό το θέμα και να εφαρμόσουμε τις συστάσεις που έχουν γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Εάν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τότε το τόπος εργασίας θα είναι ασφαλέστερος για τους ε, εργαζομένους και θα δώσουμε στον κόσμο την αξιοπρέπεια που ανέφερε ο Πάπας. Αξιοπρέπεια σε όλους τους εργαζομένους Ευρώπης. Ένα λεπτό, κυρία Κουμπούλα Ευχαριστώ. Η στρατηγική ε, μέχρι το 2012 ε, λειτουργήσε. Και είχαμε τις τρίμενες απουσίες από τον τόπο εργασία που είχαν μειωθεί περίπου κατά 30%. Τώρα έχουμε τη νέα στρατηγική, έχουμε το νέο στρατηγικό πλαίσιο που υπευλήθη. Ε, ξέρουμε ότι στόχος είναι να επεκταθούν οι, οι καριέρες και να συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι αργότερα. Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια στον τόπο εργασία. Είναι θέμα ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε να το υποτιμούμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρακτικά ε, πώ θα δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο. Α ελπίσουμε ότι θα είναι δραστήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα καλύψει ευρύτερο πεδίο ε, εξετάζοντας ε, τις συνομιλίες TTIP και όσους ενδιαφέρονται για την ε, ασφάλεια και υγεία στον τόπο εργασίας. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα κάνετε στην πράξη για όλα αυτά μετά από τη στρατηγική και με το 2012. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Έχουμε πέντε άτομα στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. έχουν, ζητήσει, έχουν ζητήσει περισσότερο το λόγο, αλλά θα επιτρέψω μόνο σε πέντε ομιλητές για ένα λεπτό και στη συνέχεια θα μιλήσει η Επίτροπος κυρία Τίσεν. Καταρχήν ο κύριος ε, Πόλτσακ από το ΕΛΚ, ο κύριος Ζάνη από τους Σοσιαλιστές, ο κύριος Μαριάς από το ECR, ο κύριος Λόβας για την ΚΟΕ, και η κυρία Μοβάη για το εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων. Ο κύριος Πότσα καταρχήν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω να αναφερθώ σε τι για να, να θέσω μια άλλη πτυχή του θέματος. Η εμπιστοσύνη μπορεί να μειώσει τους κινδύνους των εργατικών ατυχημάτων. Ε, η παρούσα κατάσταση έχει οδηγήσει σε μια υπερβολική ρύθμιση στον χώρο εργασίας. Εγώ βεβαίως ε, λυπούμαι για το κάθε θύμα, αλλά η υπερβολική νομοθεσία θα μπορούσε να μειώσει την ανταγωνιστικότητα και να αυξήσει το κόστος. Ο συνάδελφος κύριος Μάν νομίζω είπε το ίδιο πράγμα. Χρειαζόμαστε ασφαλώς μια νέα νομοθεσία, ούτω ώστε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, αλλά θα πρέπει η νέα αυτή νομοθεσία να είναι διαφανής όσο και συνεκτική. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη δική της προσέγγιση. Ο κύριος ένα για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπάθησα να διανευνήσω ήδη στο παρελθόν και τον Ιούλιο αυτού του έτους έθεσα μία ερώτηση στην Επιτροπή. Η απάντηση που έλαβα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω. Ε, μιλάμε για 24 οδηγίες σε αυτό το χώρο. Ωστόσο, η μεταφορά αυτών των οδηγιών εναπόκειται στις χώρες μέλη καθώς και η διενέργεια των ελέγχων σε σχέση με την εφαρμογή. Πιστεύω ότι η Επιτροπή στο χώρο αυτό χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη των ενδεδειγμένων εργαλείων. Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την υγεία και τις συνθήκες ασφάλειας, θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει δράση, αλλά και το Κοινοβούλιο το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν απασχολεί μόνο σήμερα την κοινωνία, να απασχολεί εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα έχει μια διάσταση ανθρώπινη, διότι η υγεία είναι σημαντικό κεφαλαιόδες αγαθό για τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχει διάσταση οικονομική, διότι εφόσον δεν τηρείται η νομοθεσία η οποία έχει επιβληθεί δίνεται την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο σε διάφορες επιχειρήσεις να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό να βρίσκουν την ευκαιρία να έχουν χαμηλότερα κόστη και βεβαίως όταν δεν τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία δημιουργούνται και αυξημένα κόστη στο ίδιο το υγειονομικό σύστημα των κρατών μελών. και αυτό είναι σημαντικό πρέπει να το λάβουμε υπόψη ιδίως στις χώρες οι οποίες έχουν υποστεί ένα χτύπημα της πολιτικής τους λόγω των μνημονίων και της πολιτικής η οποία έχει εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επισφάλεια στην εργασία και ο αποκλεισμό των συνδικάτων από τι αποφάσει που αφορούν την κλιματική υγεία και ασφάλεια είναι παράγοντε κινδύνου που η Κομισιόν δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη παρά την ε, μια αναλογική καταστροφή ε, τέτοιων ε, επαγγελμάτων έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει αυτή η τάση αν δεν ενισχυθεί η αντιπροσώπευση των εργατών στα συνδικάτα. Επίσης, λυπάμαι για την έλλειψη φιλοδοξίας της Κομισιόν μπροστά στην έλλειψη στατιστικών στοιχείων ε, και ε, στα πειράματα που γίνονται στην αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επεμβάσεις. Αντίθετα, η Κομισιόν φαίνεται αδιάφορη ε, μάλιστα και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας ε, και επιλέγει την απορρίθμιση και την αδράνεια, όπως έχει κάνει ήδη σε άλλα συναφή ζητήματα, όπως ε, στην προστασία από τα χημικά. Και πάλι εδώ αντί να βλέπουμε τη δουλειά ως ένα χώρο δικαιωμάτων, τη βλέπουμε ως κόστος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μορβάη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην Ουγγαρία υπάρχουν ε, λίγοι νομικοί οι οποίοι θα ασχολούνται με την προστασία των δικαιωμάτων ε, των εργαζομένων. Όμως ε, κάποιος από αυτούς μόλις μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό μου και αυτό το άτομο υπερασπίζεται τα θύματα των πολυεθνικών εταιριών και μου είπε ότι οι άνθρωποι φοβούνται να πάρουν αναρωτική άδεια Μάλιστα ούτε μπορούν να απομακρυνθούν για να πάνε στην τουαλέτα, δεν μπορούν να φύγουν από τις γραμμές ε, παραγωγής, πρέπει να σηκώνουν ε, βαριά άχθη, ακόμα και οι γυναίκες. Και κύριε Επίτροπε, να σας ρωτήσω τι ξέρετε για όλα αυτά και τι σκοπεύετε να κάνετε για να προστατεύσετε την Ουγγαρία και τους Ουγγρούς πολίτες από τέτοιες καταστάσεις σκλαβιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος της για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση μου δίνει την ευχαίρεια να επαναλάβω τις δεσμεύσεις μου. Θέλουμε να βελτιώσουμε συνθήκες εργασίας για τους πολίτες και θέλουμε να αφιερώσουμε την προσοχή μας στην προστασία και την υγεία στον τόπο εργασίας. Άκουσα διάφορα σημεία που υπογραμμίσατε, σημείωσα τις ανησυχίες που εκφράσατε. Δύσκολο να απαντήσω σε κάθε θέμα που θίξατε ξεχωριστά επειδή έχει περάσει και η ώρα, θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το νέο πλαίσιο. Υφίσταται το πλαίσιο, αυτό ήδη είναι κάτι καλό, είναι στοχευμένο πλαίσιο. Έτσι θα έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή των διαφορών συμφωνιών, έχουμε στόχο την πρόληψη, έχουμε σαν στόχο απαντήσεις στις δημογραφικές εξελίξεις. Κυρίως το ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια γύρανση του πληθυσμού, του ενεργού πληθυσμού. Όπως αναφέρθηκε για την ώρα κάνουμε μια εκ των υστέρων ανάλυση του κοινοτικού κεκτημένου. Έχουμε πάνω από 24 οδηγίες. Θα συνεχίσουμε το έργο αυτό, ούτω ώστε να έχουμε σφαιρικό όραμα του τι πρέπει να κάνουμε, να δούμε τι θα απορρεύσει από το νομοθετικό έργο τι έχει απορρεύσει μάλλον και να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε οργανωμένα, διαθρωμένα, ούτω ώστε να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες πολιτικές δράσεις. Στόχος είναι η βελτίωση της κατάστασης από τη συζήτηση αντελήφθην ότι θέτεται πολλά ερωτήματα όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια τον τόπο εργασία, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει η υγεία και ασφάλεια ε, των εργαζομένων να προστατεύεται στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Λιγότεροι κανόνε, συμφωνώ, αλλά όχι ει βάρο προστασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δούμε μήπω είναι δυνατό να έχουμε καλή προστασία με λιγότερε ρυθμίσει και το εγχείρημα αυτό θα πραγματοποιηθεί. Όσον αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων, πολλά συμβαίνουν παρέθεσαν κάποια από εσά αριθμητικά στοιχεία και κάθε ατύχημα είναι ένα ατύχημα παραπάνω. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά συνήγαγα από την αξιολόγηση τη πρώτη στρατηγική ότι ο αριθμό των δυστυχημάτων μειώνεται. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε επίγνωση και το εξή. Υπάρχουν νέοι κίνδυνοι οι οποίοι έχουν διαφανεί και θα πρέπει να τους προσέξουμε και να τους λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής τίθεται το θέμα του στρες που συνδέεται με την εργασία. Στο προηγούμενο πλαίσιο δώσαμε κάποια προσοχή στο θέμα και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι στο στρατηγικό πλαίσιο και ε, είναι πρόκληση και η ψυχική υγεία και το στρες. Ε, ξέρουμε όλοι μας άτομα τα οποία πάντα ε, μπορούμε να έχουμε σε επαφή μαζί τους 24 έως 24 ώρο. Έχουμε δίπλα μας όλα τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και αυτά συνεπάγονται κάποιο στρες. Και θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά εκ του σύνεγγυς. Άλλο στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στον τόπο εργασία ασκεί μια εκστρατεία τώρα, πραγματοποιεί μια εκστρατεία στους, για υγιείς τόπους εργασίας στην Ευρώπη εκστρατεία με σύνθημα ότι η υγιής εργαζόμενος αντιμετωπίζει το στρες. Ε, δεν μιλάμε μόνο ε, ε, για γενικό πλαίσιο, πρέπει να αναλυθεί και πολιτική δράση, κοινοτική δράση που πρέπει να αναλυθεί όσον αφορά την ψυχική υγεία στον τόπο εργασίας. Συντονίζεται τη δική μας Γενική Διεύθυνση όλη η προσπάθεια σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ Υπάρχει και η Γενική Διεύθυνση Υγείας βέβαια, που, που παίρνει νέο όνομα, διότι πήγε αλλού η προστασία καταναλωτών. Τέλος πάντων, θέλουμε να επιληφθούμε τη ψυχική υγεία στον τόπο εργασίας, κυρίω τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη φροντίδα. Και εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά. Ε, αναφερθήκαμε εκτενώς σήμερα και στους κινδύνους ε, από τον αμίαντο. Γνωρίζουμε ότι ο αμίαντος ε, από παλιά, εδώ και αρκετά χρόνια απαγορεύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σε διάφορα κτίρια και υπάρχουν ε, άνθρωποι που εργάζονται στις οικοδομές, που δραστηριοποιούνται στην κατεδάφιση αυτών των κτηρίων και αντιμετωπίζουν κινδύνους. Το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που πρέπει να προστατεύει τους εργαζομένους και προσθέτω ότι αυτή η νομοθεσία θα αποτελέσει ένα τμήμα του, του πλαισίου ε, των 24 οδηγιών. Αυτό που ήδη κάνουμε, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση και αποτίμηση θα δούμε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε από πολιτική σκοπιά όσον αφορά τον αμίαντο. Ο αμίαντος όμως είναι ένα σημείο που προσέχουμε η κυρία Γιούγκερ Χιούς ρώτησε τι γίνεται με τους αθλητικούς και τους αστυνομικούς. Παραδέχομαι ειλικρινά ότι δεν γνώριζα ότι αυτό το προσωπικό δεν εκαλύπτετο από την οδηγία, όμως σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτούς και θα επιληφθώ του θέματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαπίστωσα ότι σας ενδιαφέρε πολύ το θέμα. Θέλετε να κάνουμε, λάβουμε μέτρα για την υγεία και ασφάλεια ε, στον τόπο εργασία. Χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί σα. Θα πω και αυτό που είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν θα έχουμε αγαστή συνεργασία με όλου του εμπλεκόμενου φορεί και βέβαια και με του κοινωνικού εταίρου, οι οποίοι είναι οι δικοί μα εταίροι, κυρίω για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και περιμένω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Τίσεν. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Υπάρχει προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης. Αυτή η προφορική ερώτηση έχει τεθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Μαρίτα Ουλσκογκα είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το θέμα. Έχετε πέντε λεπτά, κυρία Ουλσκογκα. Η συνθήκη της Ρώμης ήδη αναφέρεται στην ε, ισότιμη μεταχείριση. Αυτό αποτελεί βασική αρχή